Η κυρία Πρόεδρος. Α, είναι Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά της ε, χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις. Οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Η ημερήσια διάταξη τώρα προβλέπει έξι προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με το Ιράν. Η περίπτωση της Ροξάνα Σαμπέρι. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες της ερώτησης, των ψηφισμάτων. Ε, ο κύριος Κέλαμ θα πάρει το λόγο πρώτος για δύο λεπτά.